Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ, καθίστε. Not many of us, but I expect the colleagues to... Δεν είμαστε πολλοί, αλλά πιστεύω ότι ανα πάσα στιγμή θα έρχονται και άλλοι συνάδελφοι. Πάντα περιμένω. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, στην τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Καταρχήν μπορούμε να συμφωνήσουμε για την ημερήσια διάταξή μας. Μάλλον ναι. Και λόγω της πίεσης χρόνου, θα σας το εξηγήσω πιο δεξοδικά αργότερα, θα σας πρότεινα να συνδυάσουμε τα σημεία 4 και 5 της ημερήσιας διάταξης δηλαδή την ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο, με τα σχόλια για τις εργασίες και την πορεία των εργασιών στην πολιτική συνοχή. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα συνδυάσουμε για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Αν συμφωνείτε με την πρότασή μου, θεωρώ ότι εγκρίνεται η σε διάταξη. Έγκριση των πρακτικών. Το σχέδιο πρακτικών της συνεδρίας 21 Μαρτίου ε, υπάρχουν στο διαδίκτυο. Οπότε συνήθω αν δεν υποβάλλετε παρατηρήσεις ή αντιρρήσει μέχρι το πέρας της συνεδρίασής μας θα θεωρηθούν ε, ότι εγκρίνονται. Έχω και μερικές ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω ότι οι συντονιστές της Επιτροπής μας ε, συνεδρίασαν στις 21 Μαρτίου μετά τη συνεδρίαση της, της Επιτροπής και οι αποφάσεις τους σας έχουν αποστελεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορούμε να τις εγκρίνουμε. Τις αποφάσεις των συντονιστών. Πολύ ωραία. Θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά της σημερινής μας συνεδρίας. Δεύτερη ανακοίνωση. Χθε το πρωί, ο κύριος Βανίστερο, η κυρία Κρέλ, ο κύριος Τζέλερ και οι υποφαινόμενοι συναντήθηκαν συζητήσαμε το γραφείο και το, το Προεδρείο συγγνώμη, και του συντονιστέ τη Επιτροπή ΚΟΤΕΡ, δηλαδή τη Επιτροπή Πολιτικής, της Πολιτικής και του Προπολογισμού τη Ένωση τη Επιτροπή των Περιφερειών, σε ένα πρόγευμα εργασία. Αντικείμενο της ε, συζήτηση ήταν ε, μια αξιολόγηση τη συνεργασία στην προηγούμενη πενταετία και διερεύνηση νέων τρόπων συνεργασία με το επόμενο Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή των Περιφερειών πρότεινε να συνοψίσουμε όλα αυτά τα θέματα σε ένα μνημόνιο που θα υποβάλλουν οι πρόεδροι των επιτροπών στα τωρινά και μελλοντικά μέλη. Και οι γραμματείες των δύο επιτροπών οριστικοποιούν ε, το έγγραφο αυτού του μνημονίου. Δεν έχουμε υπογράψει τίποτα. Πρόκειται ένα έγγραφο που ουσιαστικά κάνει μια αξιολόγηση, έναν απολογισμό της συνεργασίας των δύο επιτροπών. Στις 11 Ιουλίου η Επιτροπή Κοτέρ και η Συμμαχία για την ε, Συνοχή θα οργανώσουν συνεδρίαση για το ρόλο των συμφωνιών εταιρική σχέση ε, στη μελλοντική πολιτική συνοχή. Τα μέλη τη Επιτροπή Ρέτζι και τα τωρινά και τα μελλοντικά ε, καλούνται να λάβουν μέρος σε αυτή την συνεδρίαση. Τις λεπτομέρειες θα τις λάβετε από τη γραμματεία. Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί. Τρίτη ανακοίνωση. Μία υπενθύμηση. Έχω οργανώσει ένα μικρό κοκτέιλ κατά το τέλος της συνεδρίασής μας, εδώ στην αίθουσα. Ελπίζω να παραμείνετε να έχουμε μια σύντομη κοινωνική να παραμεινετε να εχουμε μια συντομη κοινωνικη συνέβριση για να σηματοδοτήσουμε το πέρας της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Και θα ήθελα να σε ευχηθώ να είστε καλά και καλή επιτυχία στο μέλλον, στα μελλοντικά σας σχέδια και εύχομαι και καλή επιτυχία στην ε, Μελλοντική Επιτροπή Ρέγγι και στην Επίτροπο. Καλή τύχη και καλή συνέχεια. Επίσης, τέταρτη ανακοίνωση. Να σας υπενθυμίσω, όπως είπα και στην αρχή, ότι είναι η τελευταία μας συνεδρίαση. και έχω την τιμή να προεδρεύω και έχω και κάποια προνόμια, γιατί μπορώ να λαμβάνω το λόγο όποτε θέλω. Γι' αυτό και θα κάνω αυτή την κατάχρηση του χρόνου για να ευχαριστήσω θερμά την Επίτροπο για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης θερμά όλα τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για το πολύ αξιόλογο έργο τους, ε, για το υπέροχη προσπάθειά τους, για τη μεγάλη αμέριστη υποστήριξη που μου έδειξαν και για τι κοινέ μα προσπάθειε και τι επιτυχίε μας. Λάβατε το μακροσκελή αυτό κατάλογο από τη γραμματεία. Ε, είναι ακριβώς ο κατάλογος με τις επιτυχίες μας και το κοινοβουλευτικό μας έργο στη διάρκεια της θητείας. Πολύ εντυπωσιακό κατάλογο. Ευχαριστώ θερμά τα μέλη τη Επιτροπή. Ευχαριστώ τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βοήθεια και τη συμμετοχή του. Ευχαριστώ τι υπηρεσίε του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου για την ε, βοήθεια και τη συμμετοχή του και ευχαριστώ και τις διαδοχικές προεδρίες με τις οποίες συνεργαστήκαμε με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις. Πάντως ε, αυτό που ήταν το κοινό στοιχείο ήταν ε, η πολύ αγαστή συνεργασία και η μεγάλη υποστήριξη. Να ευχαριστήσω και τους συμβούλους πολιτικής. Οι ιδιαίτερες ευχαριστίες για την ανεκτήμητη σας βοήθεια και συμπαράσταση και το έργο σας, γιατί δεν θα καταφέραμε τίποτα από όλο αυτό το μακροσκελή κατάλογο χωρί τη βοήθεια, την εμπειρογνωμοσύνη σα και τον υψηλό επαγγελματισμό σα και την εργατικότητά σα. Σα ευχαριστώ θερμότατα. Επίση, να ευχαριστήσω και τι υπηρεσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη γραμματεία μα. Θερμά ευχαριστώ στη γραμματεία για τη βοήθειά τη, για το έργο τη, για την ε, υποστηρικτική υπομονή τη, για την υπομονή σας απέναντί μου Είχαμε κάποιες απολαυστικές στιγμές και διασκεδαστικές και κάποιες περίεργες στιγμές, αλλά όλα μας βγήκαν σε καλό πάντως και ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη νομική υπηρεσία και γενικώ όλους ε, που μας βοήθησαν στο έργο μας. Και να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς, θα το επαναλάβω και στο τέλος συνεδρίασης, όπως κάνω συνήθως, αλλά να το πω από τώρα, ότι χωρίς τους διερμηνείς δεν θα είχαμε καταφέρει όλα όσα επιτελέσαμε. Γιατί μερικές φορές μπορούμε να συνεννοηθούμε με κάποιες γλώσσες, αλλά προτιμούμε να έχουμε τη βοήθεια των διερμηνών, γιατί η κατανόηση είναι καλύτερη. Θερμές ευχαριστήσεις λοιπόν και στους διερμηνείς και να ευχαριστήσω και τους καλεσμένους και τους ε, εμπειρογνώμονες που είχαμε στη διάρκεια των συνεδριάσεων. Από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από πανεπιστήμια, από διάφορους φορείς. Όλοι αυτοί μας βοήθησαν. Και έλαβαν μέρος στο έργο μας με πολύ ενεργό τρόπο κατά την τελευταία πενταετία. Και εδώ θα βάλω τελεία και θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο Κορίνα Κρέτσου. Θυμάστε την πρώτη μας ακρόαση με την Επίτροπο. Ε, μου φαίνεται σαν χθε. Και όμως δεν ήταν χθε, ήταν πριν από πέντε χρόνια. Και στο μεταξύ έχουμε επιτελέσει πολύ σημαντικό έργο και εμείς και η Επιτροπή και η Επίτροπος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Ίσκρα Μιχαήλοβα, αγαπητή Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, αγαπητά μέλη της Επιτροπής. Όντως και εγώ το θυμάμαι σαν χθε όταν πρώτο ήρθα εδώ στην Επιτροπή σας για την ακρόαση για να αναλάβω τη θέση, το χορτοφυλάκιο αυτό ε, και είναι απίστευτο ότι έχει περάσει μια πενταετία από εκείνη τη μέρα της ακρόασης μου, της πρώτης ακρόασης. Και ίσως δεν ένιωσα το πέρασμα του χρόνου, γιατί περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές και νιώθω συγκίνηση, αλλά και ταυτόχρονα χαρά. Και νομίζω ότι μπορούμε να πανηγυρίσουμε για το έργο μας, γιατί χάρη στις εργότες μας προσπάθειες και την συνεργασία μας, συνενώσαμε τις προσπάθειές μας για να μην αφήσουμε καμία περιφέρεια πίσω, κανέναν συμπολίτη μας πίσω και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό. Και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη σημερινή μέρα για να κάνουμε ένα απολογισμό του έργου μας και να δούμε τι επιτύχαμε με την κοινή μας προσπάθεια. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τις ευχαριστίες μου σε όλους σας, τις υπηρεσίες, τη διοίκηση, τους ε, διερμηνείς, στους συγητές, Ε, στις αποστολές που πραγματοποιήσαμε στις περιφέρειες και νομίζω ότι πραγματικά καταφέραμε πολλά αυτή την πενταετία. Το πρώτο μας επίτευγμα είναι ότι ε, φροντίσαμε να μην μείνει καμία περιφέρεια πίσω. Και θυμάστε το πνεύμα που επικρατούσε πριν από δύο χρόνια. Φοβόμασταν ότι δεν θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον της πολιτικής συνοχής και να έχουμε ίση κάλυψη όλων των περιφερειών. Και αυτό ήταν το μέλημά μας από την αρχή. Και νομίζω ότι καταφέραμε να το υλοποιήσουμε. Πέρασαμε και δύσκολους καιρούς το 2015 με τις μεγάλες δυσκολίες της οικονομίας στην Ελλάδα και το και λόγω τη ε, αδυναμία τη χρηματοδότηση είχαν κολλήσει πολλά προγράμματα τη πολιτική ενοχή. Πάντω, συνεργαστήκαμε με την ελληνική κυβέρνηση, είχαμε ειδικά μέτρα και ένα συγκεκριμένο προπολογισμό ώστε να μπορέσει και η Ελλάδα να ε, εκτελέσει προγράμματα υποδομών, ενέργεια, περιβάλλοντο, κοινωνικών δεξιοτήτων. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί πραγματικά ενέκρινε με πολύ ταχύ ρυθμού την αλλαγή τη νομοθεσία και συνεργαστήκαμε. Επίση, η πρωτοβουλία για να μην μείνουν ε, περιφέρειες πίσω, να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι το επίκεντρο της πολιτικής συνοχής και με αγγίζει ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Πώς να μπουν οι περιφέρειες σε ένα δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης. Και αυτό επιδιώκουμε Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορούμε να νιώθουμε υπερήφανοι για το έργο μας και τα επιτέγματά μας. Επίσης καταλήξαμε στο ίδιο συμπέρασμα για την πολιτική ε, που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τις ε, μεμονωμένες ανάγκες όπου χρειάζεται και μια προσέγγιση όχι από πάνω προς τα κάτω, αλλά αντίστροφα. Είχαμε πολλά πιλωτικά προγράμματα για τη βιομηχανική μετάβαση, για τις ε, περιφέρειες που εξαρτώνταν από τον άνθρακα και πώς θα κάνουν αυτή την ενεργειακή μετάβαση. Είχαμε αυτή την συνεργασία της στενή με τις δημόσιες αρχές και με τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών για να εφαρμοστούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να μην μείνουν πίσω οι περιφέρειες όπως είπαμε. Πολλά διδαχθήκαμε από τις προηγούμενες εμπειρίες και υποβάλαμε την πρόταση για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 και ξέρω πόσο ενδιαφέρεστε να εξασφαλίσουμε την επιβίωση αυτής της πολιτικής για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Ε, δίνουμε έμφαση στην ε, μετάβαση της οικονομίας. Αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Και η θεματική ε, συγκέντρωση των κονδυλίων. Ξεκινώντας με την πρωτοβουλία για τις περιφέρειες που θα πρέπει να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Δεν έχω χρόνο για να επισέλθω σε λεπτομέρειες της συνεργασίας μας για τις εξόχως απόκεντες περιοχές. Για παράδειγμα, είχαμε ε, στενή συνεργασία με τη Λίλιανα, με τον κύριο Μασκούρ, με τον κύριο Μαρτζή, ε, για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα υπερπόντια διαμερίσματα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τις ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές, να δείξουμε αλληλεγγύη σε περίπτωση θεομηνιών. Και έχουμε και το Ταμείο Αλληλεγγύης που στήριξε τις χώρες αυτές και τις περιφέρειες αυτές στους χαλεπούς καιρούς που πέρασαν στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και όπου είχαμε τέτοιες φυσικές καταστροφές. Και επίσης μέτρα ανακούφιση κατά τη μεταναστευτική κρίση. Δεν μπορώ να σας αφαιρώ διεξοδικά ούτε τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής. Να σας δώσω καμιά ε, νούμερα. Πάνω από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις στήριξαμε πάνω από 400.000 νέες κατά το τέλος περίοδου. Πάντως, για μένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συνεργαστεί, βρήκαμε λύσεις ε, από κοινού, στείλαμε ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα στην Ευρώπη, στην Ευρώπη μας και θεωρώ ότι το μήνυμα είναι δεν θα μείνει κανείς πίσω, καμία περιφέρεια, κανένας άνθρωπος. Και αυτό φάνηκε στην έκθεση Westphal το 2017 για τα βασικά συστατικά στοιχεία της μελλοντική πολιτικής συνοχής. Και ευχαριστώ την Κέστεν παρόλο που απουσιάζει για το έργο της αρτιότατο και ευχαριστώ και τους και οδησηγητές. Και λάβαμε υπόψη την έκθεση αυτή, την έκθεση Westphal, για τις προτάσεις μας ε, για την συνοχή μετά το 2020 και θα δείτε πολλά εδάφια της έκθεσής σας στις μελλοντικέ μας προτάσεις. Έχουμε διατηρήσει την πολιτική αυτή για όλες τις περιφέρειες με ισότιμη, πιο ισότιμη κατανομή των πόρων με βάση την ε, γνωστή μέθοδο του Βερολίνου. Ε, επικεντρωθήκαμε σε βασικές προκλήσεις της οικονομικής μετάβασης και της μετάβασης σε μια οικονομία χωρίς ε, εκπομπές άνθρακα και παρόλα αυτά στηρίζουμε τις υποδομές ε, ε, και τις ε, κοινωνικές υποδομές σε υγεία, παιδεία και δεξιότητες, χωρίς τη δική σας ενεργό συμμετοχή, χωρίς τη δική σας συμπαράσταση και συνεργασία δεν θα μπορούσαμε να, είχα, να καταφέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Και όταν βλέπω το έργο μας, ε, διαπιστώνω ότι έχουμε και άλλα επιτεύγματα. Καταρχήν, φέραμε την πολιτική αυτή πιο κοντά στους πολίτες και μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Η επικοινωνιακή μας πολιτική ήταν βασική προτεραιότητα της θητείας μου και χαίρομαι που βρήκαμε ε, κοινό παρανομαστή εδώ. Γιατί δείχνει πια και το Ευρωβαρόμετρο ότι... Ε, παλιά μόνο ένας στους τρεις πολίτες γνωρίζουν τα επιτεύγματα της ε, πολιτικής συνοχής επιτόπου. Και χαίρομαι που δεν ήμουν μου όταν προσπάθησα να φέρω ε, τους πολίτες πιο κοντά στην πολιτική αυτή. Με βοηθήσατε κι εσείς και είχαμε συμπληρωματικές προσπάθειες και με τη διαδραστική πλατφόρμα «Τι κάνει η Ευρώπη για μένα» καταφέραμε να αποδείξουμε στους πολίτες ότι η πολιτική συνοχή και τα προγράμματά της έχουν ε, απτά αποτελέσματα στις περιφέρειες. Επίσης έχουμε και την πλατφόρμα με τα ανοιχτά δεδομένα που ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ για τη μη υποστήριξατε και με την Επιτροποτά. Σε το 2017 για την ανακοίνωση για, τη για τα, τις 7 δράσεις. Είχαμε 1.700 διαβουλεύσεις για την πολιτική συνοχή στην Ευρώπη και 450.000 άνθρωποι συμμετείχαν ε, στα ερωτηματολόγια και στις ε, διαβουλεύσεις αυτές. Ήταν ε, πραγματικά εντυπωσιακό επιτεύγμα και με τον κόσμο για το τι κάνει η πολιτική συνοχή στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ και για την βοήθεια στην τοπική ανάπτυξη 1.300 τοπικές στρατη... αναπτυξιακές στρατηγικές παρουσιάσαμε, γιατί οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ε, λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και αυτό ήταν μία από τις πέντε προτεραιότητες μας για το μέλλον. Ε, η βασική προτεραιότητα η Ευρώπη κοντά στους πολίτες επιτρέπει την τοπική ανάπτυξη σε αστικές και αγροτικές περιοχές και δίνει κίνητρα για τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και της τοπικής κοινότητας προκειμένου να προωθεί ένα ε, μια αίσθηση οικειότητας με τα τοπικά προγράμματα ε, με βάση και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ και για την πρότασή σας για την διασυνοριακή συνεργασία και ευχαριστώ τον Πασκάλα Ριμό για την έκθεσή του για τη διασυνοριακή συνεργασία. Γιατί αυτή η συνεργασία είναι η πιο απτή και ορατή πτυχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματο δείχνει ότι η Ευρώπη είναι παρούσα παντού. Και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και ότι διεκπαιρώσατε αυτό το θέμα. Το ίδιο ισχύει και για τη στρατηγική και τις μακροπεριφέρειες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε και θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της στρατηγικής για τις μακροπεριφέρειες. Θέλουμε συνεχή υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο ρόλος σας ήταν πραγματικά κρίσιμος. Άλλη επιτυχία μας ήταν η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την απλούστευση και την καλύτερη εφαρμογή. Περάσαμε ώρες ολόκληρες να ακούμε τις μορφές για τις περίπλοκες διαδικασίες, τη γραφειοκρατία και όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου διαπίστωσα αμέσω ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και να κάνουμε την πολιτική συνοχή πιο φιλική προς το χρήστη, τον αποδέκτη. Και εκεί με βοηθήσατε πολύ και στον κανονισμό Omnibus ε, προτείναμε απλουστευμένες ε, λύσεις και πολλές ε, άλλες προτάσεις για να περιοριστεί η γραφειοκρατία. Και αυτό το καταφέραμε χάρη στην ενεργό συμμετοχή των εισηγητών. Ο Ενίστερ Ρόιτς, της Κωνσταντσε Γκρέλ, ευχαριστώ Λάμπερτ και να μεταφέρει σε μου και στην Κωνσταντσε. Λάμπερτ, αφήνει μια πραγματικά τεράστια παρακαταθήκη. Σε ευχαριστώ θερμά. Δεν είχαμε μόνο εύκολες στιγμές, αλλά τα καταφέρουμε και πιστεύω ότι θα κρατήσουμε τη φιλία μας. Η πείρα σας ήταν πολύτιμη και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμότατα, Λάμπερτ. Φυσικά έχω θερμές ευχαριστίες και για την Ίσκρα, αλλά όλοι σας βοηθήσατε γιατί έχετε γνώση της κατάστασης επιτόπου και γι' αυτό στις επίσημες αλλά και τις άτυπες συναντήσεις μας με βοηθήσατε να διαμορφώσω μια γνώμη και με παροτρύνατε να λάβω υπόψη την εμπειρία σας. Μαζί με τον κανονισμό Omnibus ξεκινήσαμε τις ε, προετοιμασίες για μια πλούστερη πολιτική συνοχή μετά το 2020. Και όπως είπα, η ενεργός συμμετοχή ήταν πολύ χρήσιμη. Προτίσα, προτείναμε 80 μέτρα πλούστευσης, ε, εξορθολογισμό του προγραμματισμού, ε, πλούστερη και ταχύτερη εφαρμογή και τα προγράμματα έτσι θα, μπορούσαν, θα επικεντρωθούν περισσότερο στη βοήθεια των αποδεκτών και στην ε, εφαρμογή αποτελεσμάτων. Πολύ συγκεκριμένα από τα επιτεύγματα λοιπόν της πολιτικής συνοχής, οπότε μπορούμε να επιστρέψουμε στις πατρίδες μας και να πούμε ότι δώσαμε μάχη για μια πολιτική πιο κοντά στους πολίτες, για απλούστευση, να μην μείνει καμία περιφέρεια πίσω, για καλύτερη εφαρμογή. Οπότε όλο αυτό το αξιόλογο έργο θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και να ευχαριστήσω την κυρία Ίσκρα Μιχάηλοβα, την Πρόεδρο, για τις για τους χρονοβόρους τριμερείς διαλόγους. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε για τον νέο κανονισμό και τον προϋπολογισμό του κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Θα μείνει για το επόμενο κοινοβούλιο. Πάντως, μακάρι να είχαμε καταφέρει να συμφωνήσουμε πριν τις ευρωεκλογέ, ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή από την 1η Πρώτη του 2021 για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Παρ' όλα αυτά ελπίζω να προλάβουμε και να καταλήξουμε στη συμφωνία πριν τα τέλη του έτους. Γιατί χρειαζόμαστε προγράμματα που θα πρέπει να τρέχουν και να χρηματοδοτηθούν και γι' αυτό το νομοθετικό πακέτο θα πρέπει να υιοθετηθεί το συντομότερο δυνατό. Όπως είπα μόνο εγκόμια έχω και επένος για την Επιτροπή σας, γιατί άοκνα εργαστήκατε ε, για να διαμορφώσουμε την πολιτική συνοχή μετά το 2020 ιδιαίτερε ευχαριστίε προ την πρόεδρο αλλά και στου ηγητέ, την κυρία Κρέλ, τον κύριο Νοβάκοφ, τον κύριο Κοτσολίνο, τον κύριο Αριμό, τον κύριο Βαν Μίλτεμπουργκ. Εργαστήκατε ε, σκληρά για να προετοιμάσετε τι εκθέσει και να ετοιμαστείτε για τι διαπραγματεύσει. Εσείς κάνατε ό,τι μπορούσατε, κάνατε τα δύνατα δύνατα, αλλά δυστυχώ το Συμβούλιο ανέκοψε αυτή τη διαδικασία. Πάντως ε, έχουμε πολλά κοινά σημεία στις θέσεις μας και τους τριμερείς διαλόγους αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Χαίρομαι και για το επικοδομητικό πνεύμα που πριτάνευσε στους τριμερείς διαλόγους. Με απογοήτευσε παρόλα αυτά η έλλειψη πρόοδου και λυπάμαι που δεν καταλήξαμε σε συμφωνία γιατί μας μπλόκαρε το Συμβούλιο. Πάντως ελπίζω το επόμενο Κοινοβούλιο να συνεχίσει τη δική σας πορεία και να εκμεταλλευτεί το, την παρακαταθήκη που αφήνατε. Εν πάση περιπτώσει αυτά έχει ζωή. Ο χρόνος περνάει γρήγορα. Είναι η τελευταία φορά που είμαι εδώ μπροστά σας ως Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής. Ελπίζω όμως να επανέλθω ως Ευρωβουλευτής ίσως στην επόμενη θητεία. Πάντως χαίρομαι για τα επιτέγματά μας. Είμαι υπερήφανη για τα επιτέγματά μας. Τα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα. Αυτή ήταν σημαντικότατη πρόκληση εξόχως απόκεντρες περιοχές, αστικά κέντρα, περιοχές εξαρτημένες από το άνθρακα και πώς θα πραγματοποιήσουν την βιομηχανική τους μετάβαση. Δεν θα μπορούσα να είχα ευχηθεί πιο καλούς εταίρους και συνεργάτες. Ήταν τιμή μου που συνεργαστήκαμε και σας εύχομαι καλή τύχη στο μέλλον, καλή συνέχεια και όπου και αν ξανασυναντηθούμε μπορούμε να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τους συμπολίτε μας και για τις περιφέρειές μας. Εδώ κανονικά θα έλεγα ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αυτή τη φορά όμως δεν θα πω μόνο ευχαριστώ για την προσοχή σας, αλλά ευχαριστώ για όλα. Η πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε. Πραγματικά χαρά και τιμή για μας να συζητούμε μαζί σας, ως συνήθως κάθε φορά που ήρθατε δηλαδή στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και όπως πρότεινα να συνδυάσουμε δύο πράγματα, δηλαδή την συζήτηση με την Επιτροπό και την συζήτηση του έργου μας και την πρόοδο στην πολιτική συνοχή μέχρι τώρα αλλά και τα προβλεπόμενα για το μέλλον, να σας δώσω λίγα νούμερα, τα οποία περιλαμβάνονται και στην επισκόπηση που έχει συντάξει η γραμματεία και σας την έχει διαβιβάσει. Αλλά πιθανώς ακόμα να μην τα έχετε διαβάσει με όλες τις λεπτομέρειες. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι για τις τρεις πρώτες νομοθετικές προτάσεις για τη μελλοντική πολιτική συνοχή, δηλαδή CPR, η e RDF και Interreg και Ταμείο Συνοχής, συν τον μηχανισμό για τα ευρωπαϊκά σύνορα, που ήταν οι τέσσερι μεγάλοι φάκελοι για του οποίου ήταν υπεύθυνη η Επιτροπή Περιφερειακής ανάπτυξη. και μπορέσαμε να επιτύχουμε ε, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια. Πολύ σημαντικό και με ικανοποίηση άκουσα χθε τη συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειών ότι οι περιφέρειες εκτιμούν το έργο μας, κατανοούν την δυσκολία που είχαμε για να φτάσουμε σε συμφωνία μεταξύ ημών και του Συμβουλίου. Η πρώτη ανάγνωση όμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο εκτιμούν ιδιαίτερο τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειών και κατανοούν τη δυσκολία του έργου μας και μάλιστα μας συνεχάρισαν. Δεύτερο, είχαμε 16 άλλες νομοθετικές διαδικασίες οι οποίες πέρασαν από την ε, ε, Επιτροπή μας, ορισμένες πολύ γρήγορα λόγω διαδικασία κατεπίγοντο που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, εμείς δείξαμε κατανόηση και επιτύχαμε να περάσουν γρήγορα. Επίσης, συντάξαμε 25 νομοθετικές νομοδοτήσει για άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπές και αυτό δείχνει ότι η συνεργασία με τι άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ ήταν θετική και καλή. Και ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη εργασία τη Επιτροπή μα σε τούτη εδώ τη θητεία ήταν η πολύ καλή συνεργασία με τι άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και το υψηλό επίπεδο κατανόηση. Σπανίω ε, ε, βρεθήκαμε σε σύγκρουση ενδιαφερόντων με τι άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και εν πάση περιπτώσει και σε αυτέ τι συγκρούσει εμεί κερδίσαμε. Ε, επιτύχαμε. Επίσης, 29 μη νομοθετικές προτάσεις ή μάλλον εκθέσεις όπου περιλάβαμε τις θέσεις μας και σε έπτα εκθέσεις εφαρμογής. Κάτι που δεν είναι πολύ δημοφιλές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί άλλες επιτροπές έχουν λιγότερο, μικρότερους αριθμούς τέτοιου είδους, τέτοιου είδους εκθέσεων. Εμείς είχαμε όμως και είχε ενδιαφέρον. Ο κύριος Μάτο άνοιξε μάλιστα τον δρόμο στις implementing αυτές εκθέσεις και 15 αντιπροσωπείες των μελών μας για να δουν την εφαρμογή, την εκτέλεση δηλαδή της πολιτικής συνοχής επιτόπου. Άρα έχουμε πράγματα, πράγματι πολλά να συζητήσουμε. Θα σταματήσω τώρα, θα δώσω τον λόγο στα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, αρχίζοντας βέβαια από τους συντονιστές. Τρεις βρίσκονται στην αίθουσα. Ας αρχίσουμε με τον κύριο Βανίστελροϊ του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ. αντιλαμβάνεστε ότι ε, επειδή την τελευταία ομιλία καθενό την κρατάνε στο μυαλό του οι περισσότεροι, περισσότερο από την πρώτη, θα προσέξω το τι θα πω. Όταν είδα την υποψηφιότητα της ε, κυρίας Επιτρόπου και την είδα να κυκλοφορεί στους διαδρόμους κλπ. Ε, της είπα πάντοτε να προσέχει να προσέχει ορισμένα θέματα γιατί ιδίως για την ψηφιοποίηση που είναι σημαντική και τώρα να σας πω το εξή. Έγινε η ακρόαση βεβαίως της κυρίας Κρέτου μετά, ΕΕ και κάποιο μαγικό έγινε, διότι οι πολιτικέ ομάδε βέβαια θέτουν ερωτήσεις Και βέβαια μπαίνει κάποια προτεραιότητα. Εγώ ανεπίσημα είχα θέσει τι ερωτήσει. και τελικώ έτσι, επειδή είχα θέσει πολλές φορές τι ερωτήσει, δεν ήθεσα εκείνη τη φορά. Και όμω απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή απάντησε η Επίτροπο στην ακρόασή τη, θέλω να πω, χωρί καν να έχω θέσει την ερώτηση. Ήταν όμω ερώτηση την οποία είχα θέσει πολλέ φορέ πιο πριν. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι καμιά φορά ε, ε, επιτυγχάνουμε όταν έχουμε κάνει διαρκή προσπάθεια. Και αν δείτε τι επιτύχαμε εν τέλει. Εγώ προέρχομαι μια χώρα που είναι καθαρός φορεύς. Και να σας εξηγήσω και τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι με επικρίνουν διαρκώ στη δουλειά που κάνω εδώ. Διότι πάντοτε εμφανίζομαι προβολικά θετικό για την πολιτική συνοχή. Η πολιτική συνοχή όμω είναι η συγκολητική ουσία που κρατεί τις περιφέρειες, ε, τις πόλεις, ε, τους δήμους, τις κοινότητες, όλα αυτά τα, τα, κρατεί, τα, συγκρατεί μαζί. Και στην Ολλανδία ο υπουργό μας των οικονομικών μου λέει «Ε, αυτά μου κοστίζουν λεφτά. Και ποιο είναι το αντάλλαγμα. Κάνεις και τα υπολόγισα και του είπα ότι δεν, μπορεί να, δεν μπορείς να έχεις ακριβώς ε, τα ακριβή ανταλλάγματα. Αλλά ε, αυτή είναι η δική του αντίληψη. Πάντως θεωρώ ότι ε, επιτύχαμε ένα μικρό θαύμα. Και αυτό που είπε και η ίδια η κυρία Επίτροπος για όλες τις περιφέρειες που εξυγχρονίστηκαν προσεγγίζοντας και τους πολίτες. Ε, απορροφά βέβαια αυτό το 1 τρίτο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διάφορα πράγματα τις ε, τελευταίες αυτές μέρες της παρούσης θητείας. Δεν θέλω βέβαια να στρέφω τα μάτια μου μόνο προς τα πίσω. Όμως το, στην ανεπίσημη διάσκεψη κορυφής εχθές για την περιφερειακή συνεργασία με τους Κινέζους και αν δείτε τι λένε αυτοί. Μας ρώτησαν πώς τα καταφέρατε ε, ε, κάνατε διεύρυνση με 12 νέε χώρε ε, και μάλιστα πολλέ από αυτέ τι φτωχέ. Περάσατε από μια κρίση και καταφέρατε να ανακάμψετε. Πώ τα καταφέρατε, με, τις μεγάλες, με τη μεγάλη ανάπτυξη βέβαια των παράκτιων περιοχών, αλλά αυτοί που, έχουν οι Κινέζοι δηλαδή, και βέβαια με την τεράστια ενδοχώρα. Έχουν ένα τεράστιο πληθυσμό, έχουν ε, εκτάσει. εκτάσεις. Αν τα εξετάζει κανεί βέβαια από την απόσταση αυτή για το τι κάνουμε εμείς εδώ για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Βλέπουν ότι η πολιτική συνοχή δεν είναι μια ασπιρίνη, είναι στην πραγματικότητα πολιτική πρόληψη για να αποφευθούν πολλά στραβά που μπορούν να συμβούν στην κοινή μας Ευρώπη. Και ακριβώς όπως είπε η πρόεδρός μας κυρία Μιχαήλοβα, είχαμε δηλαδή και πολλούς αγώνες μέσα στη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να περάσουμε τις θέσεις μας. Αν δούμε δηλαδή ότι τα διαθωτικά ταμεία στηρίζουν προγράμματα, διαθωτικά ταμεία που στηρίζουν προγράμματα, δεν ξεκινά από την Οικονομική Επιτροπή, εδώ γίνεται. Εμείς λάβαμε τη θέση αυτή διότι είχαμε θέση. Και ε, αυτό είναι που θέλω να πω όταν θα μπορέσω να απευθυνθώ στο επόμενο ε, κοινοβούλιο που θα έρθει, στους επόμενους ευρωβουλευτές. Μην χάσετε τις ευκαιρίες που έχετε. Να εξυγχρονιστείτε, να κάνετε όλες τις αναγκαίες ε, τροποποιήσεις και προσαρμογές για να αντιμετωπίσετε και επερχόμενα προβλήματα, μεταναστευτικό, ε, προσφυγικό, σεισμοί, mm. παρακμή των αστικών κέντρων. Για λογαριασμό του Λαϊκού Κόμματος λοιπόν μπορώ να πω ότι για μένα η συγκίνηση είναι μεγάλη όταν σκέπτομαι τι έγινε για παράδειγμα στις περιοχές της Υπέθρου. Και ε, συμφωνία για τα ε, εφή χωριά, όπως κάναμε και με το πρόγραμμα για το ΕΦΗΕΣ Άμστερνταμ. Μιλώντας πάντως για τις θέσεις αυτές, γιατί έχουμε την πέμπτη προτεραιότητα στο νέο κανονισμό μας, δηλαδή προσέγγιση στους πολίτες. Χρειάζονται οι επόμενοι ευρωβουλευτές να έχουν πολύ ισχυρότερες θέσεις γι' αυτό, για το τι μπορούν να συνεισφέρουν για τη σταθερότητα του μέλλοντος της Ευρώπης, να μην πέσουν στην παγίδα του εθνικισμού και σε αυτά τα προβολικά συντηρητικά λαϊκιστικά πράγματα που στρέφονται κατά της Ευρώπης. και να έχουν και άμεση γραμμή επαφής με την επόμενη, με την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στο πιλωτικό πρόγραμμα επίσης συνέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συμμετοχή τριών επιτρόπων για την ε, μετακίνηση προς πιο βιώσιμες ενέργειες και βεβαίως για την φροντίδα υγείας. Οι άνθρωποι γυράσκουν. Θα χρειαστεί ένα άλλο κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο που πρέπει να το δούμε. Δεν θα γίνει από μόνο του. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Βλέποντας την Ευρώπη απ' έξω Βλέπετε και τώρα του ΟΣΑ την έκθεση του 2012 που μιλεί για τρία πράγματα. Ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση, τεχνολογικές αλλαγές, δημογραφικές αλλαγές, αστικοποίηση, γύρανση του πληθυσμού, μεταναστευτικό και αλλαγή του κλίματος. η δουλειά που κάναμε είναι προς αυτές τις κατευθύνσεις. Και εδώ ευχαριστώ όλους και όλους τους συναδέλφους για την συνεργασία και βεβαίως όλο το προσωπικό που κατέστησε δυνατή αυτή τη συνεργασία. Νομίζω ότι η περίοδος αυτή ήταν πραγματικά, έχει, ο απολογισμός είναι θετικός. Σας ευχαριστώ κύριε Βανίστερ Ρόι. Um, Van Ευχαριστώ. Κύριε Βαν Βίλτεμπεργκ, έχετε εσεί το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε, ε, αγαπητή Επίτροπε, Αναφερθήκαμε στην αρχή της θητεία ε, και της συνεργασίας όταν ήσασταν εδώ ως υποψήφια επίτροπο. Αν χθε μα φαίνεται, ενώ ήταν πριν από πέντε χρόνια και απαριθμίσατε όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει. Κάναμε σπουδαίο έργο νομίζω και με τις δικές σας προτάσεις για εξοχρονισμό της πολιτικής συνοχής ώστε να εξασφαλίσουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη την στήριξη των επενδύσεων, την αλληλεγγύη, ε, Νομίζω μπορούμε να, συγχα... να σας συγχαρούμε λοιπόν. Αλλά μοιράζομαι μαζί σας ε, την απογοήτευσή σας όσον αφορά το νομοθετικό έργο προς το τέλος της εντολής. Ε, δεν υπήρξε μεγάλη πρόοδος για τη CPR, ε, τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Παρότι είχαμε εμείς τη βούληση, το Συμβούλιο εργάστηκε πάνω στην Ευρωπαϊκή Δαφική Συνεργασία, το Ταμείο Συνοχής το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το κανονισμό όμως για το Αναπτυξιακό Ταμείο δεν υπήρξε πρόοδος επιτόπου πραγματική και αυτό με απογοητεύει όπως και εσά, γιατί θα έπρεπε να περιμέναμε από την Ρουμανική Προεδρία να έχει ανάμεσα στις προτεραιότητες της την πολιτική συνοχής. Περισσότερο από ό,τι υπόλοιποι. Υπάρχουν ακόμα όμως λίγες ελπίδες γιατί αύριο θα είστε στη Βουκουρέστη για να συζητήσετε σε μια άτυπη συνεδρίαση με τους υπουργού την ε, απάντηση, την ε, ε, θέση για την συνοχή. Ποιο θα είναι το βασικό σας θέμα ε, και μήνυμα, γιατί εκεί θα μιλήσετε για τα κονδύλια, για το ευρωπαϊκό ξε... Ε, εξάμεινο. Ε, υπάρχουν πάνω κάτω οι θέσεις της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου και στο επίπεδο της Κορεπέρ υπάρχουν κάποιες θέσεις στο Συμβούλιο που δεν κατευθύνονται πάντοτε προς τη κατεύθυνση των δικών σας προτάσεων. Έχετε δει τι εγκρίναμε στην Ολομέλεια για το Ταμείο Συνοχής πριν από δύο εβδομάδες. Άρα λοιπόν, τι θα προσπαθήσετε εσείς να διαβιβάσετε στους υπουργούς ως μήνυμα κλειδί. Μια από τις ανησυχίες μου είναι ότι αν δείτε τις θέσεις του Συμβουλίου ας πούμε, για τον κανονισμό του, ε, του Ταμείου Συνοχής θέλουν να βάλουν ε, το σημείο 5 στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Πιστεύω πως είναι κρίσιμο για την Ευρώπη. Αν θέλει να είναι πρωτοπόρος όσον αφορά την καινοτομία και αν δεν θέλει να χάσει τον αγώνα κόντρα στους Αμερικανούς και τους Κινέζους, να διατηρήσουμε αρκετά χρήματα για, την διαπεριφερεια... για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις ε, για την καινοτομία. Είναι ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα προσφυλές, γιατί βεβαίως η περιφερειακή πολιτική δεν αφορά μόνο την αλληλεγγύη, δεν αφορά μόνο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, αλλά ε, θέλει να καταστήσει την Ευρώπη ισχυρότερη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, επίσης, πώς από κοινού θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό το συστατικό να, να, εκπέσει, να μην είναι ούτε στο Ταμείο Συνοχής, ούτε στο Ταμείο περιφερικής Ανάπτυξης. Ε, αυτό κάπως με ανησυχεί. Οπότε το θέμα είναι, θα είναι και αυτό θέμα της ε, αυρινής σας συζήτησης, αύριο. Θα είναι κομμάτι της προσπάθειας της Επιτροπής να μείνουμε στη δική σας πρόταση. Και μετά έχω και μια πιο πρακτική ερώτηση και ο Λάμπερς αναφέρθηκε στην αστική ατζέντα. Είναι σημαντικό να υπάρξει ε, μια, ένα επίσημο ανακοινοθέν προς το Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά τα πορίσματα των ε, στατικικών θεματικών εταιρικών σχέσεων. Να μην ξεχνάμε δηλαδή αυτή την ατζέντα και να επιστήσουμε την προσοχή του επόμενου Κοινοβουλίου στον απολογισμό αυτής της διαδικασία. Τέλος, θα, θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία και στο εγγύς μέλλον. Εσείς είστε υποψήφιο, έχετε καλό βέβαια βιογραφικό, ε, ε, αλλά θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και της ομάδας μου του Άλντε για την καλή μας συνεργασία στο πέρασμα των πέντε ετών και ακόμα και αν φαίνεται σαν χθες, ε, το αυριανό ε, το αύριο θα έρθει και αυτό πολύ γρήγορα και σας εύχομαι, όπως είπα, καλή επιτυχία και στην αυριανή σας συνεδρίαση με τους υπουργού ε, που είναι αρμόδιοι για την περιφερειακή πολιτική. Κρατήστε σκληρή στάση εκ μέρους της Κομισιόν και εκ μέρους του Κοινοβουλίου, ώστε να λειτουργήσει η ε, πολιτική συνοχής και στο μέλλον και να εξυγχρονιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, thank you, Mr. Van Miltenburg. Thank you. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που μας θυμήσατε την αυριανή συνεδρία στο Βουκουρέστι να σας ενημερώσω ότι θα έχουμε και δικούς μας εκπροσώπους εκεί. Ο κύριος Ομαρζέ θα, ως πρώτος αντιπρόεδρος της, Επιτροπής, ε, της Περιφερειακής Επιτροπής και ο κύριος Ζέλερ θα εκπροσωπήσουν την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σε αυτό ε, το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών και θα παρουσιάσουν τα επιτεύγματα της Επιτροπής μας και τις θέσεις μας. Θα έχουμε λοιπόν λόγο και εμείς εκεί αύριο. Κυρία Νταμάτο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Προέδρε και ευχαριστώ Επίτροπε που είστε εδώ στην τελευταία μας ε, συνεδρίαση της Επιτροπής. Εγώ ήθελα να προσπαθήσω να συνοψίσω, να κάνω ένα απολογισμό για τα τελευταία πέντε έτη της ε, θητείας, ε, για τα μέτρα που έχουν ε, εγκριθεί, αλλά και για το τι μας περιμένει είτε σαν βουλευτές είτε σαν πολίτες. Εν γέννη, όταν εγώ και το κίνημα από το Πέντε Αστέρων φτάσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο, βρισκόμασταν ενώπιον ενός όρους λιτότητας και εκ μέρους σας υπήρχε μεγάλη δυσπιστία απέναντι σε αυτό το νέο κίνημα που για πρώτη φορά ερχόταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο, και όλα τα ηθάκελοι επί των οποίων αρχίσαμε να ε, δουλεύουμε ε, είχαν ε, ξεκινήσει με ένα είδος θρησκείας που βασιζόταν στην, τυφλή, στο τυφλό δόγμα της λιτότητας. Εμείς λέγαμε από το 12 ότι έπρεπε να ακυρωθεί το, ε, το θέμα αυτό και τελικά η πλειοψηφία ε, του Ευρωκοινοβουλίου μας έδωσε δίκαιο. γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη, ο αγώνας για το κλίμα, η ιδεολογική ε, προσπάθεια και η ασφάλεια των σεισμικών περιοχών δεν μπορούν να διακινδυνεύονται, δεν μπορεί δηλαδή να περιορίζει τις διορθωτικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις μια χώρα όταν τις επιβάλλονται εκ των άνω και μάλιστα εφόσον πρόκειται για μια πολιτική λιτότητα η οποία έχει αποτύχει και ο ίδιο ο πρόεδρο Γιούνκερ το είπε πρόσφατα. Και όταν πρόκειται για την εφαρμογή τέτοιων αρχών για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Για μα είναι φρικτό λοιπόν που η Κομισιόν προσπάθησε και συνέχισε να προσπαθεί να προτείνει αυτό το μέσο. Εύχομαι ότι στην επόμενη θητεία θα, θα μπλοκαριστεί η μακροοικονομική ερεσιμότητα οι επιτυχίε για την καταπολέμηση τη λιτότητα δεν σταματούν εδώ στην Ιταλία και στις Βρυξέλλες. Διάφοροι πολιτικοί ε, ηθήνοντες έχουν επιτεθεί και συνεχίζουν να ε, ε, μάχονται κατά ε, υπέρ μάλλον του εισοδήματο, του μήνυμου εισοδήματο. Στην Ιταλία το έχουμε ήδη εγκαταστήσει. Μα λέγανε ότι ήταν τρέλα, όμω ε, στην Ιταλία λειτουργεί και μάλιστα για, με βάση το κοινωνικό ταμείο 21-27 είχε προβλεφθεί η δυνατότητα να ε, ληφθούν τέτοιου είδου μέτρα όπω το ε, μήνυμου εισόδημα για τον πολίτη. Βλέπετε, Επίτροπε, όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούσα να καταλάβω πώς η δική μου αντιπροσωπεία ιδιαίτερα ε, εδώ έχει διακριθεί και έχει δείξει υπευθυνότητα. Οπότε έχουμε δείξει ότι δεν παρακολουθούμε τους ε, διάφορους μύθους, ότι προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών που εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν κρατηθεί σε απόσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Μάλιστα συνεργαστήκαμε επικοδομητικά για τους τρεις κανονισμούς, ας πούμε το Interreg, το, το κανονισμός για τις κοινέ διατάξεις. Και είμαι ευτυχής που μπόρεσα εγώ προσωπικά να συμβάλλω, αλλά και ως αντιπροσωπεία για να εγκριθούν κανόνες που είναι ένα σημείο εκείνης εξαιρετικό για το επόμενο κοινοβούλιο. Και αυτό είναι καρπός ε, της συνεργασίας όλων, όπως είπαν και οι συνάδελφοι και η πρόεδρός μας. Για το Ίντερεγκ, για παράδειγμα, χάρη στην ε, συνεργασία αυτή εδώ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, ε, μπορέσαμε να παρέμβουμε στα διάφορα κρίσιμα σημεία. Και στο νέο κανονισμό καταφέραμε να αναβάλουμε την θαλάσσια δυσυνοριακή συνεργασία και το βάλαμε στο πρώτο άξονα. Τι άλλο να πω, ε, και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις περιείχε διάφορα κρίσιμα πράγματα, το νησιν 2 για αναφέρω που είναι ιδιαίτερα τιμωρητικό για τις, τα διάφορες μας περιφέρειες ή ακόμα η μεταφορά προς μέσα άμεσης διαχείρισης και η μείωση του, του ποσοστού συγχρηματοδότησης. Όμως η ολοκληρωμένη και υπερψηφισμένη πρόταση στο Ευρωκοινοβούλιο πέρα από την, ε, ε, τις Μα μικροοικονομικέ ερεσιμότητες είχε και περιλαμβάνει και επιτυχίες. Δηλαδή αύξηση από 322 στα 378 δις, ε, αναγνωρίζοντας έτσι συμμαχίες συνοχής για την ανάπτυξη και την εξέλιξη και την ανάπτυξη των διαφόρων μας περιφερειών, πώς ε, ε, εισήχθη ο κανόνας νησιν 3 και αυξήθηκαν, αυξήθηκαν οι επενδύσεις. Είναι ένα βήμα μπροστά. Βεβαίως το πρώτο βήμα μόνο γιατί ε, Είχαμε πολύ σημαντικά θέματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ζήτημα για το οποίο μίλησα πριν, το αυθινόπορο, ε, θα πρέπει τελείως να ακυρωθεί και το Κοινοβούλιο να προωθήσει ε, την θέση της Ολομέλειας. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή λοιπόν και θα υπερασπιζόμαστε αυτά τα αποτελέσματα. Τέλος, για το ε, το Κοινοβούλιο έχει τροποποιήσει το ποσοστό θεματικής συγκέντρωσης. Βασιζόμαστε στην οικοδόμηση των τριών επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών. Θέλω να κλείσω με ένα χαμόγελο και μια θετική νότα. Πιστεύω πως και η Κομισιόν ε, θα, και η Επίτροπος μάλλον θα το δεχτεί και θα χαρεί για το νέο άρθρο 6. Αυτό που σταματά την χρήση των στερεών καυσίμων, των καυσίμων, θυμίζω ότι πριν από δύο εβδομάδες η Ολομέλη έδειξε θάρρος, ίσως και περισσότερο, από την Κομισιόν και έδειξε μεγαλύτερη διορατικότητα λέ, αποφεύγοντας το χρήση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για να ε, χρηματοδοτηθούν οι ε, πηγές ε, ορυκτών καυσίμων. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την Πρόεδρό μας, της υπηρεσίας του Κοινοβουλίου και να ευχαριστήσω και την Κοινοβουλευτική Ομάδα και τον πολιτικό σύμβουλο μας, τον Ανδρέα Πικόλ, που είναι πάντοτε διαθέσιμος. Ελπίζω ελπίζω στην επόμενη θητεία με κάποιο τρόπο ακόμα και οι συνάδελφοι που δεν θα είναι υποψήφοι και, αλλά που έχουν συμβάλει με την εμπειρία τους θα μπορούν πια ως πολίτες και ως σύμβουλοι μας να συμβάλλουν. Γιατί το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να παγιώσουμε τα καλά αποτελέσματα αυτής της θητείας και να επαναλάβουμε και περισσότερο. Ευχαριστώ. Thank you, Ms. Uh, colleagues. Ευχαριστώ κύριε Δαμάτο. Ποιο άλλο θα ήθελε το λόγο, ο κύριο Σουλάκ. Σα um, Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ και ακούσαν αρκετά, από... έχουν σκυλοβαρεθεί τους Βρετανούς τις τελευταίες εβδομάδες. Εγώ δύο χρόνια έχω ε, ε, που συμμετέχω σε αυτήν την Επιτροπή, αλλά εκτιμώ την καλή εργασία και τις καλές προθέσεις της Επιτροπής και της Επιτρόπου. Ίσως ε, να επιστρέψω για, λίγο, για, για ένα σύντομο διάστημα, αλλά σίγουρα όχι αρκετό. Ναι, είμαι υποψήφιος. Ε, συγγνώμη παιδιά, θα με ξαναδείτε. Αλλά μπορεί το Halloween να φύγουμε πια. Ίσως εκεί να είναι και πιο κατάλληλη περίοδος. Σε αυτό το σύντομο λοιπόν χρονικό διάστημα, ίσως να μην πρέπει να σας κουράσω με ερωτήσεις και με θέματα που μπορεί να απασχολήσουν τα επόμενα πέντε χρόνια. Πάντως εξ ονόματος των Βρετανών συντηρητικών και της αντιπροσωπείας του ECR που είμαι εκπρόσωπος της, δεν βλέπω άλλου συναδέλφου εδώ. Θα ήθελα στην Επιτροπή, την Επίτροπο να την ευχαριστήσω για την εργασία τη και για την Πρόεδρο για την εξαιρετική Προεδρία. Τέλος, ε, να πω κάτι που πολλοί έχουν πει και πολλοί θα έχουν ακούσει και παλιότερα. Το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει όχι γιατί εχθρεύεται την Ευρώπη. Οι περισσότεροι δεν εχθρευόμαστε την Ευρώπη. Εγώ σίγουρα όχι. Αυτό αφορά το προβληματισμό μας σε σχέση με ολόκληρο το project ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε, ε, ξέρουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον και στις μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες καλή επιτυχία για το μέλλον. Thank Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι, ευχαριστώ βεβαίως και ολόκληρη την αντιπροσωπεία της ε, συντηρητική κοινοβουλευτική ε, κοινοβουλευτικής σας που στάθηκε επικοδομητικά κοντά μας σε όλα τα θέματα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πολύ καλημέρα σας. Θα ήθελα και εγώ μια κοινή τελευταία μας συνεδρίαση και επειδή θα σταματήσω το πολιτική δραστηριότητα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πολύ ευγενικό αλλά και αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο προεδρεύατε στις συνεδριάσεις μας. Και ευχαριστώ και τους βοηθούς μας, τους υπαλλήλους, τους συναδέλφους, τους διερμηνείς και ε, να συμφωνήσω και εγώ με τα εγκομιαστικά σχόλια που ακούστηκαν για τον συντονιστή της ομάδας μου, τον κύριο Βανίστε Ρόι. Πραγματικά έμαθα πολλά μαζί του και από την πλούσια πείρα του. Οι 24 χρόνια ήμουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ήμουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε είχα μία άποψη για την πολιτική συνοχή, την πολιτική συνοχής και αφιέρνω τον ελεύθερο χρόνο μου και τα Σαββατοκύριακα σε επαφέ με νέους από την πατρίδα μου. Και αυτό το μήνυμα θα ήθελα να συμμεταφέρω. Ε, όποιος έζησε την Πορτογαλία και πριν και μετά την ένταξη είναι ανενδίαστα υπέρμαχος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάπειρος φιλοευρωπαίος πατρίδα μου δεν θα ήταν τίποτα σήμερα χωρίς την πολιτική συνοχή. Είναι αδιανόητη ε, και τεράστια η πρόοδος που επιτύχαμε χάρη στην ένταξη. Επίσης, για τον πέμπτο στόχο στο επόμενο πρόγραμμα, καλό θα ήταν να τον τονίσουμε, για να γνωρίσουν οι πολίτες τι κάνει η Ευρώπη για αυτούς. Γιατί ένα από τα βασικά προβλήματα της Ευρώπης ε, είναι ότι η πολίτες που είναι βασικοί αποδέκτες της πολιτικής συνοχής μερικές φορές το αγνοούν. Αγνοούν τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς. Και αυτό φταίνε μερικές φορές οι αρμόδιοι για την επικοινωνία που δεν καταφέρουν να προβάλλουν τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής και έτσι δεν αναγνωρίζεται ούτε ο ρόλος των χώρων, των χωρών συνεισφορέων αλλά ούτε και τα ωφέλη για, τις, για τους αποδέκτες. Ε, όντως ε, πέρασαν σε μια πνοή τα πέντε χρόνια. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η πενταετία αλλιώς ε, χαρακτηρίζει τους άνδρες και τις γυναίκες. Οι άνδρες ε, γερνάνε κατά πέντε χρόνια, ενώ οι γυναίκες ξανανιώνουν, γίνονται πέντε χρόνια νεότερες. Έτσι λέμε εμείς στην Πορτογαλία, ότι ο χρόνος περνάει μόνο για τους άνδρες. Κύριε Πόλτσακ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στην Επίτροπο την κυρία Κρέτσου για το έργο της. Και θα ήθελα να την ευχαριστήσω για το ρόλο που έπαιξε στην ενίσχυση της πολιτικής συνοχής. Αναλάβατε τα καθήκοντά σας σε δύσκολους καιρούς. Περάσαμε πολλές κρίσεις. Την κρίση με την Ουκρανία, την κρίση της Ελλάδας κρίσεις που επηρέασαν την πολιτική συνοχή. Επίσης είχαμε τη μεταναστευτική κρίση, μετά το Brexit και άλλες κρίσεις που έπληξαν την Ευρώπη. Χαίρομαι πάντως που η πολιτική συνοχής έμεινε αλόβητη παρά τις κρίσεις και εξακολουθεί να έχει κέριο ρόλο και σημασία. Χαίρομαι λοιπόν που καταφέραμε να κάνουμε αγώνα και να διαφυλάξουμε την πολιτική συνοχή και το μείζωνα ρόλο της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για αυτόν τον κοινό αγώνα και τα επιτεύγματα, να ευχαριστήσω τον συντονιστή μας και κυρίως την πρόεδρό μας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ροντρίγκε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερος την Επίτροπό μας για τη συνεργασία που είχαμε, τους συναδέλφους, τους υπαλλήλου και τα εύσημα στην Πρόεδρο, που πραγματικά με υποδειγματικό τρόπο προείδρευσε. Μέσα αυτή την πενταετία είχαμε και κάποιες στιγμές έντασης, αλλά είχαμε πολύ περισσότερες ε, επικοδομητικές στιγμές παρά τεταμένες. και χαίρομαι ε, γιατί όταν ε, ήταν λάβουμε ε, σημαντικές αποφάσεις και για την Πορτογαλία και την Ισπανία είχαμε ενιαία στάση και φωνή και στην Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και την Επίτροπο για την προσοχή που έδωσαν στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Σας ευχαριστώ θερμά. Ή για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και περιφέρειες. Επίσης προσπαθήσαμε να μην τις αφήσουμε πίσω και στο μέλλον θα πρέπει να προστατεύσουμε την πολιτική συνοχής και θα τα καταφέρουμε όχι μόνο δίνοντας έμφαση στα οικονομικά ζητήματα και στα επενδυτικά που έχουν φυσικά τη σημασία τους, αλλά να τονίσουμε την συμβολή της πολιτικής συνοχής στην ενίσχυση της Ευρώπης και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Και μερικές φορές ε, οι εθνικές κυβερνήσεις ε, σφετερίζονται τις δικές μας επιτυχίες και τα δικά μας κατορθώματα. Θα πρέπει λοιπόν στον τρόπο που επικοινωνούμε με τους Ευρωπαίους πολίτες να τονίζουμε το τι προσφέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω γιατί ε, είμαι καθηγήτρια και ερευνήτρια και θα πρέπει λοιπόν να να προσπαθήσουμε να διαπαιδαγωγήσουμε όχι μόνο τους νέους, αλλά και τους υπόλοιπους πολίτες που αγνοούν το έργο μας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνιακή μας πολιτική. Θα πρέπει επίσης ε, να απλουστεύσουμε και στην πολιτική συνοχή, αλλά και στις άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης τον τρόπο επικοινωνίας μας με τους πολίτες. Η πολιτική συνοχή ε, είναι η φωνή των περιφερειών. Οπότε, αν δεν καταφέρουμε να μεταφέρουμε ε, το έργο της και την αντίληψη του έργου της πολιτικής συνοχής της Περιφέρειας είναι σαν να έχουμε αποτύχει, ενώ έχουμε κάνει τόσα θετικά αυτή την πενταετία που μας πέρασε. Και κάτι άλλο. Έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολες εκλογές. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί να πούμε ότι ε, υπάρχει έντονος λαϊκισμός ή δημαγωγία. Θα πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας και τον αγώνα μας κατά της δημαγωγίας και του λαϊκισμού. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη και την αγάπη των Ευρωπαίων πολιτών προς την Ευρώπη. Αυτή ε, θα πρέπει να είναι η δύναμή μας στις επόμενες ευρωεκλογές. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Ροντρίγκες και ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια. Ο κύριος Ομαρτζή. Ευχαριστώ. Όταν έχουμε μια τελευταία συνεδρίαση επικρατεί ένας πιο ε, πανηγυρικός τόνος. Ε, δυστυχώς ο χρόνος περνάει ε, και εμείς τον ακολουθούμε. Ο χρόνος περνάει σίγουρα, αλλά παρόλα αυτά κάναμε πολλά σε αυτή την πενταετία. Και ευχαριστώ την πρόεδρο ε, της Επιτροπής μας, την κυρία Μιχαήλοβα, για την κομψότητα με την οποία διαχειρίστηκε την Προεδρία. Ε, έδειξε μεγάλη λοιπόν κομψότητα στην άσκηση της Προεδρίας και μεγάλη διαθεσιμότητα και συνεργασία μαζί μας. Θερμά ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, για 26 χρόνια διατέλεσα δήμαρχος και θα σας ε, εξομολογηθώ κάτι. Ε, μερικές φορές ε, επέκρινα και εγώ την πολιτική συνοχής ως δήμαρχος. Αλλά όταν ήρθα εδώ και έγινε ευρωβουλευτής, διαπίστωσα ιδίως όμως... Όμαση πόσο σημαντική είναι η πολιτική συνοχή για τι περιφέρειες, για τα διάφορα εδάφη και κυρίω για τα υπερπόντια εδάφη και τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Όντω κάνατε πάρα πολλά και μάλιστα σε πολύ δύσκολου καιρού και με μεγάλε αντικσότητε. Αλλά είναι αδιαφυσβήτητο ότι δείξατε μεγάλη βούληση ευήκονους αφού γραστήκατε τις ε, ανάγκες και τις, τα αιτήματα των ε, εξόχως απόκεντρων περιοχών και των υπερπόντιων διαμερισμάτων. Και σας ευχαριστώ εκ μέρους των συναδέλφων. Τρεις είμαστε από υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας, έχουμε άλλους συναδέλφους από τις εξόχως τις περιοχές και νομίζω ότι πολύ πρόοδο σημειώσαμε. Και αν έχουμε φανεί πρόοδο στην ανάπτυξη των ε, εδαφών και των περιφερειών μας, αυτό οφείλεται και σε εσά. Το 30% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξυπηρετεί την ανάπτυξη των εδαφών και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά είχαμε πολύ ωραίες νίκες και επιτεύγματα. Για τη φορολογία για το Ρούμι, για παράδειγμα, για τις εξόχους τις περιοχές και για την Αλία είχαμε μια μεγάλη επιτυχία. και η ανανέωση της αλληλίας για παραλληλευτικά δι, δι, ε, ήδη ε, βελτιώθηκε. Μας βοηθήσατε σε πολλά μέτωπα ε, για την ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Μόνοι μας δεν θα τα καταφέρναμε χωρίς τη δική σας βοήθεια. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που πραγματικά ήταν πολύ δεκτικοί και ανοιχτοί να μας βοηθήσουν και να προωθήσουν τα θέματά μας. Εγώ μετά από 42 χρόνια πολιτικού βίου εγκαταλείπω την πολιτική σκηνή και χαίρομαι που θα ολοκληρώσω την πολιτική μου σταδιοδρομία ως Ευρωβουλευτής. Η θητεία μου ήταν πολύ επικοδομητική. Έμαθα πολλά από εσά. Έμαθα πόσο χρήσιμη και απαραίτητη είναι η Ευρώπη. Και η Ευρώπη που τόσο πολύ μας εξυπηρετεί και μας βοηθά, δυστυχώς είναι παρεξηγημένη και άγνωστη για πολλούς συναδέλφους. Θέλουμε μια Ευρώπη, Ευρώπη πιο πολιτική, πιο κοντά στον κόσμο, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί έχουμε εμείς ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη εμάς. Σας ευχαριστώ. Thank you so much, Mr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μασκούρα. Ο κύριος Χάτμαν και μετά εσείς. Κύριε Χέτμαν. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τα δικά μου εγκόμια και τις εγκάρδιες ευχαριστίες των συναδέλφων. Πραγματικά σας ευχαριστώ για την εξαιρετική εργασία και συνεργασία που είχαμε στην, ε, περιοχή, ε, στην Επιτροπή. Από την πρώτη στιγμή ήταν πολύ ευχάριστη η συνεργασία με την Επίτροπο, με την Πρόεδρο, με τους συναδέλφους, τα μέλη της Επιτροπής. Συγχαρητήρια και στο συντονιστή μας, τον κύριο Βανίστερ Ρόι. Του είμαι ευγνώμων γιατί έχω μάθει πάρα πολλά από αυτόν από τη γνώση του, από την εμπειρία του. Αλλά ευχαριστώ και τους άλλους συναδέλφους με τους οποίους συνεργαστήκαμε ε, πολύ στενά ε, για την πολιτική αυτή και για την πολιτική συνοχή μετά το 2020. Καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες για να σφυριλατήσουμε αυτή την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι αυτή η ενίσχυση της αλληλεγγύης είναι ίσως η πιο ανεκτήμητη συνεισφορά και η μεγαλύτερη και σημαντικότερη μας παρακαταθήκη. Γιατί δυστυχώς πολλοί εγωισμοί ε, εμφανίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε ε, περιφέρειες με άνισο επίπεδο ανάπτυξης. Προσπαθήσαμε να μην μείνει καμία ε, περιφέρεια πίσω, να κερδίσει το χαμένο έδαφος, αλλά λαμβάνουμε υπόψη ακόμη και τις προηγμένες ε, περιφέρειες, γιατί και αυτές έχουν προβλήματα. Θα ήθελα, κυρία Επίτροπε, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία. Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για την ε, μεγάλη χάρη με την οποία ασκήσατε και κομψότητα την Προεδρία να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πολύ επικοδομητική και ουσιαστική συζήτηση και συνεργασία που είχαμε και να, να επαναλάβω την ευχαριστία μου, τις ευχαριστίες μου προς τον κύριο Πανίστερα με τον οποίο έμαθα πάρα πολλά και ελπίζω τη γνώση που αποκόμισα από τη συνεργασία μας να την μεταφέρω και στις υπόλοιπε μου ε, δράσεις και στη συνέχεια της ζωής μου. Νομίζω ότι Όλοι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το έργο που επιτελέσαμε την πενταετία που μας πέρασε. Γνωρίζω ότι το έργο αυτό την χάνει ιδιαίτερη εκτίμηση σε επίπεδο ε, δήμων, κοινοτήτων και περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκ μέρους των περιφερειών και της Πολωνίας θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, ο κύριος Γκάμπελη. Ο κύριος Γκάμπελη, ευχαριστώ πολύ. Ένα χρόνο ήμουν εδώ. Αντικατέστησα τον Νίλσον, που δυστυχώς απεβίωσε προέτους και όμως είχε δουλέψει καλά εδώ. Και εδώ, αλλά και στην Βόρεια Σουηδία. Και εγώ έχω να πω καλά πράγματα και να πω ότι έμαθα πολλά για την πολύ και καλή δουλειά που κάνετε εδώ και που κάναμε και μαζί και είδα και τη σημασία της πολιτικής συνοχής, της περιφερειακής συνοχής στην πράξη και πόσο σημαντικό είναι να κρατηθεί η Ευρώπη ενωμένη σε περίοδους δύσκολες. Θα πω λοιπόν και εξ ονόματος της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που προσωπώ μόνος μου σήμερα εδώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Επίτροπο και καλή επιτυχία στο μέλλον, καθώς επίσης θα ευχαριστήσω την κυρία Πρόεδρο και ε, τους υπολείπους, προσωπικό κλπ. Και συνεχίστε να εργάζεστε για την βελτίωση της Ευρώπης. Μένει ο κύριος Βέρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ είναι σωστό να λάβω τον λόγο παρόλο που είμαι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής σας. Ωστόσο ήταν σημαντικά τα πράγματα που διδάχθηκα εδώ για την πολιτική μου καριέρα. Ευχαριστώ τον Βανίστερ Ροϊδίο ιδιαίτερος για την υποστήριξη που μου προσέφερε. Πραγματικά μας έσπροχνε διαρκώς ε, σε μια ε, ας πούμε πιο έντονη δέσμευση και εμπλοκή. Συνεργαστήκαμε με θαυμάσιο τρόπο και με πολύ ευχάριστο τρόπο, χωρίς βαθιές πολιτικές διαφωνίες. Και αυτό οφείλεται και σε εσά, κυρία Πρόεδρε, που καταβάλατε μεγάλη προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί αυτό. Η κοινοβουλευτική μας επιτροπή θα μπορούσε να ονομάζεται και Επιτροπή Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, διότι η αλληλεγγύη είναι άλλωστε η βάση, το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κατανομή των αναπτυξιακών κονδυλίων στις περιοχές εκείνες και περιφέρειες της Ευρώπης που τα χρειάζονται αποτελεί έκφραση μεγάλης αλληλεγγύης την οποία προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ως κοινοβουλευτικό σώμα βεβαίω συμβάλαμε σημαντικά. Γι' αυτό και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που μπόρεσα να αποτελέσω μέλος της μεγάλης αυτής οικογένειας στην ε, λίγουσα τώρα κοινοβουλευτική θητεία. Και καλή επιτυχία στο μέλλον, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ βεβαίω και το προσωπικό τη Επιτροπή. Εγώ έχω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλους για τα πολύ καλά σας λόγια. Τώρα θα επιστρέψω το μικρόφωνο στην κυρία Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους σας για τα καλά σας λόγια, για τις ευχάριστες αναμνήσεις που μοιραστήκαμε για όσα συνέβησαν από την αρχή της ε, θητείας, για την ευφυή εξειδίκευση και άλλα πράγματα που καταφέραμε μαζί και όπως είπατε θα μπορούσε να είχαν γίνει πολύ περισσότερα. Θα προσπαθήσω εγώ με τη σειρά μου να απαντήσω σύντομα σε κάποιες από τις ερωτήσεις που κάνατε, διότι κατά τα λοιπά συνεργαστήκαμε και ελπίζω θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ώστε να επιτύχουμε και άλλα πράγματα. Όπως είπα στην ομιλία μου πριν, κύριε Βαν Μίλτενμπουργκ, ε, μοιράζομαι την απογοήτευσή σας, ε, διότι δεν επιτεύχθη συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογέ, που ήταν η μεγάλη φιλοδοξία του Πρόεδρου Γιούνκερ, αλλά και δική μου. Και ε, ήταν και πάρα πολύ σημαντική για τις χώρες μέλη και για τις περιφέρειες. Ελπίζω ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος για την έγκριση του νομοθετικού πακέτου δεν κατέστη δυνατό. Ελπίζω ωστόσο να επιτευχθεί η συμφωνία μέχρι τέλους του έτους. Και ένα από τα μηνύματα μου αύριο στο Συμβούλιο, στο Βουκουρέστι δηλαδή, θα είναι να ενθαρρύνω τις χώρες μέλη να προχωρήσουν με τις διαπραγματεύσεις για, το, για την νομοθετική δέσμη μέτρων, ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν άμεσα οι τριμερείς διάλογοι. Με το νέο που θα προκύψει από τις ευρωεκλογές, δηλαδή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για μας, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Δεν έφταιγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που, άρχισε, που άργησε να αρχίσει ο, ο ε, τριμερής διάλογος, διότι την πρόταση μας την είχαμε έτοιμη είναι σημαντικό να αρχίσουμε τις επίσημες συζητήσεις για τον προγραμματισμό επιτόπου. Εάν οι τριμερείς διάλογοι δεν γίνουν, δεν αρχίσουν στην αρχή της επόμενης προγραμματικής περίοδου, πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσουμε να, ολοκληρώσουμε τον προγραμματισμό για την επόμενη περίοδο ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να πληρώνουμε τιμολόγια από την 1η Ιανουαρίου 2020, όταν θα εγκριθεί το νομοθετικό πακέτο. Οι ανταλλαγές απόψεων και συζητήσεις θα συνεχιστούν. Εγώ αγωνίζομαι πέρα της πρότασης της Κομισιόν, που είναι ξεκάθαρη. Αλλά βέβαια, είμαστε και έτοιμοι και έτοιμες να συζητήσουμε οποιαδήποτε πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από την πλευρά των χωρών μελών. Ελπίζω ότι έτσι απαντώ στην κυρία Νταμάτο και στον κύριο Μίλτενμπορκ. Η πρότασή μας είναι τώρα στα χέρια του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που είναι οι συνομοθέτες. Αλλά ευχαρίστως να συμβάλλουμε δίνοντας τις αναγκαίες εξηγήσει και κάνοντας προτάσεις ώστε να ε, διευκολυνθεί η προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους κράτους των περιφερειών σας. Τους περιφερειάρχες σας. Κάνουν σπουδαία πράγματα στην Επιτροπή Περιφερειών. Και είναι αναγκαία η συμμαχία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπή Περιφερειών για την υλοποίηση των προτάσεών μας. Είπα για την επικοινωνία και άλλα πράγματα που θέτουμε εδώ, ότι πρέπει να φτάσουμε στα αυτιά και του τελευταίου πολίτη. Η Ευρώπη, το ευρωπαϊκό project δεν αφορά μόνο τις Βρυξέλλες, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αφορά κάθε χώρα μέλος, κάθε περιφέρεια, κάθε δήμο και κοινότητα και κάθε πολίτη. Αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να επισκεφτώ στο δυνατόν περισσότερες περιφέρειες, ευρωπαϊκά έργα, να αντιληφθούν οι πολίτες ότι αυτός ο εξυγχρονισμός του τάδε νοσοκομείου, ε, η κατασκευή του τάδε αυτοκινητοδρόμου, προέρχεται από την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσα ίσως να είχα επιτύχει περισσότερα, αλλά Έπρεπε να είμαι και εδώ. Έπρεπε να έρχομαι να βλέπω και το κοινοβούλιο. Έκανα λοιπόν ό,τι μπορούσα με τον τρόπο μου και σας ευχαριστώ όλες και όλους, όπως είπα, για τα καλά σας λόγια και όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, επιτύχαμε πολλά, αλλά το πιο σημαντικό που επέτυχε η Επιτροπή περιφερειακής αναπτύξεως είναι τελικώ η κληρονομιά που θα παραδώσετε στους επόμενους και αποτελεί καλή βάση για την επόμενη Επιτροπή Περιφερειακής ε, Ανάπτυξης που θα αναλάβει τα ενία μετά τις ευρωεκλογέ. Δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο, σας ευχαριστώ και πάλι και ελπίζω να σας ξαναδώ μετά τις εκλογές. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή τύχη και σε εσά και στις οικογένειές σας και στις χώρες σας. Ευχαριστώ. Thank you, Commissioner. Σας ευχαριστούμε Επίτροπε. Εδώ ολοκληρώνονται οι συζητήσεις μας. Ε, ολοκληρώσαμε την σημερινή ημερήσια διάταξη και έχω το αγαπημένο μου σημείο. Διάφορα. Υπάρχει κάτι στα διάφορα κύριε Βανιστερόη. Οι επιτροπές μας είναι ενδιαφέρουσες γιατί είναι πολύ ζωντανε. Έχω μια ερώτηση. Τα πιλωτικά μας πέρασαν. Όλα, ναι. Ίσως να έχουμε την απάντηση. Από τη δική μου πλευρά, ναι. Όλα τα πιλωτικά έχουν μεταφερθεί έχουν σταλεί στην Επιτροπή Προπολογισμού και στην Κομισιόν. Αν η Κομισιόν θέλει τώρα να πει κάτι, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, ξέχασα εγώ τι έχει γίνει. Έχουμε εδώ τους εκπροσώπους των υπηρεσιών μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω εξάλλου όλους για, για τη σκληρή δουλειά και την αγαστή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Να ευχαριστήσω και τις πολιτικές ομάδες και τις γραμματείες. Είναι καθήκον μου να ευχαριστήσω και το επιτελείο μου στην Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ. So, we, we concluded any other business. Κάτι άλλο. Εγώ όταν θα λέω τα διάφορα θα θυμάμαι πάντα τον κύριο Φαναριστερόη. Σας ευχαριστώ όλους. Θέλω συνεδρίασης και συνεχίζουμε με μια σύντομη εκδήλωση για ένα ποτηράκι κρασί εδώ. Εδώ στην αίθουσα αυτή. Και επίσης μαζί με τον, την Επίτροπο Θα κάνουμε μια σύντομη συνέντευξη έξω από την αίθουσα. Σας ευχαριστώ όλους.